Ε, σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τα εξής θέματα. Ε, τον κανονισμό σχετικά με το κοινοτικό σήμα και ε, τα τέλη που καταβάλλονται στο Γραφείο Εναρμόνισης. Επίσης, την, οδηγία, την αναδιατύπωση της οδηγίας που συγκλίνει τις νομοθεσίες των κρατών μελών για τα σήματα. Στη σημερινή